φάρμακα που σώζουν ζωές στην Ευρώπη. Και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβετε το λόγο η Επίτροπος Χέντιγκορτ. Περιμένουμε μερικά λεπτά μόνο. Κύριε Λάιχτφριτ, εσείς θα συνοδεύσετε τον Επίτροπο που αποχωρεί και μπορεί να ξεκινήσει κύριε Χέντιγκορτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι κυρίε και κύριοι εκ μέρου ε, του συναδέλφου Επιτροπού Μπόρς ήθελα να πω ότι ε, συμμερίζεται τις ανησυχίες σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την διάθεση νέων ιατρικών φαρμάκων ε, νέων φαρμάκων και τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περιθαλψή. Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να δώσει ε, την απαραίτητη μέρημνα και φροντίδα. Έχουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση του Απριλίου του 2014 για ένα αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα υγείας, για ανθεκτικά και αποτελεσματικά συστήματα υγείας, δηλαδή μια αποτελεσματική πρόσβαση στα συστήματα παροχής ε, υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως λέγαμε, καλύτερη συνεργασία, διαφάνεια, συντονισμό για να αποτραπούν οι εσδήποτε αντίξουες ε, συνθήκες μπορεί να προκύψουν από τα εθνικά συστήματα υγείας σε σχέση με την προσβασιμότητα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας τον Ιούνιο μια αντιπροσωπεία και συγκεκριμένα η Γαλλική επισήμανε το ιδιαίτερο ζήτημα της ε, νέας ε, αγωγής για την υπατήτηδα C που είχε λάβει έγκριση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέφρασε την ε, ανησυχία της σε σχέση με τη δυνατότητα πρόσβαση του είδους θεραπεία. Αύριο ειδικοί, των, ε, ε, ειδικοί εκπρόσωποι και πυρογνώμες των κρατών μελών ε, θα συζητήσουν τα θέματα αυτά. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Συμβουλίου και των Αρμοδίων Αρχών σε σχέση με την τιμολόγηση και την αποζημίωση των αγωγών. Και βεβαίως το ζήτημα της τιμής, το πόσο δηλαδή οικονομικά είναι ανεκτό, ανεκτή η τιμή ενός φαρμάκου και μιας αγωγής, δεν περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της υποτίθετας γάμα. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στις πρωτοβουλίες ε, για το προσεχές ε, ανεπίσημο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για την καινοτόμο υγεία που έχει προαναγγελθεί από την Ιταλική Προεδρία την επόμενη εβδομάδα. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί μια συζήτηση για την οικονομική διάσταση της καινοτόμου ιατρικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα θα βοηθήσει και θα επιταχύνει τη διαδικασία για πιο καλά και πιο αποτελεσματικά φάρμακα. Η Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Νομοθεσία περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία που εξασφαλίζουν ε, έγκαιρη και πρώιμη πρόσβαση ε, σε φάρμακα για ασθενείς που έχουν ε, ιδιαίτερου χαρακτήρα οι απρόβλεπτες ιατρικές ανάγκες και ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολύ σπάνιες και επικίνδυνες για την υγεία ε, ασθένειες. 106 καινοτόμες ε, θεραπείες και αγωγές έχουν εγκριθεί εν προκειμένου, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμιά εξουσία να προσδιορίσει τιμολόγιο για αυτές τις αγωγές. Αυτό είναι κάτι που ανήκει στο κάθε κράτος μέλος χωριστά ως αρμοδιότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ορίσουμε ανώτατο όριο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει την αρρωγή της όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, παραδείγματι ως προς την ε, τιμολογιακή πολιτική για να αποτρέψει αρνητικές συνέπειες ως προς την προσβασιμότητα στα φάρμακα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας θα ήταν να εξετάσουμε ένα σύστημα κοινού μηχανισμού προμηθειών έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές από πλευρά της φαρμακευτικής μηχανίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χέντεγκαρτ. Και τώρα ο κύριος Μικολάσικ για δύο μισή λεπτά. Äh, Ευχαριστώ πρόεδρε, ναι, κύριε Επιτρόπε συνάδελφοι. Αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να μας ε, βοηθήσει ε, να ε, μελετήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα τους ασθενείς, ε, ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με το πώς θα σώσουμε ζωές. Η βελτίωση της πρόσβασης ε, σε φάρμακα που σώζουν ζωές ε, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και ιδιαίτερα ανθρώπους σαν και εμένα που είμαστε γιατροί. Εγώ δούλευα ε, παλιότερα σε νοσοκομεία, στο, στην κλινική που ε, δεχόμασταν ασθενείς με πολύ σοβαρές ασθένειες και θα έπρεπε εμείς να τους σώσουμε τη ζωή. Ε, είμαι λοιπόν, μου είναι λοιπόν οικείο το θέμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που ε, έχουμε διαθέσιμα ε, για να προωθήσουμε τέτοιου είδους φάρμακα, ε, η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και συχνά οι ψηλές τιμές των φαρμάκων αντικατοπτρίζουν την έρευνα που απαιτείται προκειμένου να παραχθεί, να το φάρμακο αυτό. Οι φάρμακοβιομηχανίες ε, ε πολύ συχνά ε, έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν πολύ ψηλές τιμές. Ε, από το 2000 2009 η ιατρική φαρμακευτική διαπάνη μάλλον αυξήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 76%. Τεράστια αύξηση. Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γυράσκει βέβαια και οι τιμές των καινούριων φαρμάκων ε, αυξάνονται όλο και περισσότερο. Τα σημαντικά φάρμακα όμως θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε λογικές τιμές στους ασθενείς που τα χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μικολάου. Κυρία Μπορζάν για 1,5 λεπτό. Ε, Κύριε Πρόεδρε, η ιατρική πρόεδρος προσφέρει αποτελεσματικά αλλά και ακριβά πολύ συχνά φάρμακα. Όταν εμφανίζονται λοιπόν φάρμακα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σε 100% θεραπεία, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιατρός ο οποίος μπορεί να σταθμίσει ε, την υγεία του ασθενούς έναντι της εξοικονόμησης ε, πόρων. Αλλά αν πρέπει να μιλήσουμε για την τιμή ενός ε, φαρμάκου, φαρμάκου που μπορεί παραδείγματι να θεραπεύει και την υπατήτηδα γάμα, θα πρέπει να δούμε τι θα σήμαινε το αντίστροφο. Δηλαδή τι θα σήμαινε αν ένας ασθενής δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει αυτή την αγωγή. Εάν έπρεπε να πάει να κάνει ενδεχομένως μεταμόσχευση ύπατος, εάν έπρεπε να λείψει τόσες μέρες από τη δουλειά του, εάν εν τέλει έχανε και τη ζωή του ακόμη. Όλα αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα τα οποία μας ανησυχούν ε, σημαίνουν ότι πρέπει να έχουμε, ότι χρειαζόμαστε ένα σοβαρό, ένα καλό αποτελεσματικό σύστημα υγείας και χρειαζόμαστε πόρους για τη χρηματοδότηση των ε, φαρμάκων και θεραπείων, ιδιαίτερα όταν μπορούν να συμβάλλουν σε μια ε, πλήρη θεραπεία. Θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε το ζήτημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την προστασία αυτών και τη διάρκεια αυτών σε σχέση με τα φάρμακα. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι η Ιταλική Προεδρία προσπαθεί να συζητήσει όμως υπό τον ε, τομέα των ε, εμπορικών συναλλαγών, στο εμπορικό δίκαιο δηλαδή και όχι στο τομέα της δημόσιας υγείας που πραγματικά αξίζει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πορζάν. Η κυρία Φων Στόρχ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε όλοι υποστηρίζουμε την ε, προστασία της ανθρώπινης ζωής και γι' αυτό και την ως το δυνατόν ευρύτερη διάδοση και πρόσβαση σε φάρμακα μπορεί να σώσουν ζωές. Σε σχέση όμως με αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις, ε, στην έρευνα σε εμβριακά βλαστοκύτταρα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 18 Οκτωβρίου του 2011 έλαβε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, έδωσε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση και διευκρίνησε ότι η ανθρώπινη ζωή ξεκινάει ε, η ανθρώπινη ζωή που θέλουμε να προστατέψουμε ξεκινάει όταν συναντιέται το οάριο με το σπερματοζωάριο. Ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει με την ένωση οαρίου και σπερματοζωαρίου. Με βάση αυτήν την ε, νομολογία θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε μέσον το οποίο θα μπορούσε να σημάνει παρέμβαση, χειρισμό ή και καταστροφή ανθρώπινου όντως. Έχουμε μια πρωτοβουλία πολιτών που ονομάζεται One of Us, ένας από εμά και που έχει ζητήσει την απαγόρευση της ε, έρευνας με, τα, με εμβριακά βλαστοκύτταρα. 1,8 εκατομμύρια πολίτες υπέγραψαν και υποστήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως υπό τους χριστιανοδημοκράτες έχει παρά το γεγονός ότι 1,8 εκατομμύρια πολίτες υπέγραψαν αυτή την πρωτοβουλία πολιτών αγνοήσει τις φωνές τους και ε, παραγνωρίζει το γεγονός ότι καταστρέφεται ανθρώπινη ζωή με την έρευνα αυτή στα ε, εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φωνστόρχ. κυρία Μπετσέρα ε, κυρία Επιτροπέ, άκουσα με προσδοκία και με ενδιαφέρον την άποψη της Κομισιόν. Ε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το χρόνο μου προκειμένου να προβάλλω την ανάγκη να εξυπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον. Ε, πότε μπορούμε μια παθολογική κατάσταση να την καταστήσουμε, ε, να, να θεωρήσουμε ότι ε, είναι σοβαρή. 130 εκατομμύρια άτομα έχουν πληγεί από την... 130.000 άτομα έχουν πληγεί από την πατήτιδα C. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει θεραπεία. Κοστίζει παραπάνω 50.000 ευρώ κατά άτομο την τιμή αυτή την καθόρισε η εταιρεία που παρήγαγε το φάρμακο με καθαρά εμπορικά κριτήρια. Τι θα γίνει, πάλι θα αναζητήσουμε προσχήματα ε, και δικαιολογίες για την αδράνειά μας. Πάλι θα υποστούμε το ζυγό των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 31 της διακήρυξης της ε, Ντόχα ε, του ΠΟΕ. Τα κρατημέλη μπορούν να το κάνουν. Ε, για λόγους δημόσιας υγείας μπορούν να ε, παραβούν την, ε, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να παράγουν γενώσιμο φάρμακο στη θέση του πρωτότυπου. Μπορούν να κάνουν από κοινού δημόσιες προμήθειες. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος αγοράζει γενώσιμο φάρμακο από την Ινδία 100 φορές πιο φτηνά το πρωτότυπο. Άλλες ε, ανάπτυξη χώρες θα ε, επωφεληθούν από την απόφαση της Ινδίας να παράγει ε, γενώσιμα φάρμακα κατά παράβαση των διπλωμάτων βρεσιτεχνίας. Αν εμείς καταφέραμε να βάλουμε όρια στο roaming στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν θα έπρεπε να μπορούμε να θέτουμε όρια σε τέτοιου είδους πρακτικές για να σώσουμε εκατομμύρια ζωέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέτσερα Μπαστερετσέα και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Χρυσόγονος. Το πρόβλημα της υπερκοστολόγησης των φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες με σκοπό να αποκομίσουν υπερκέρδη σε βάρος της υγείας των πολιτών και σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων είναι υπαρκτό αλλά δεν είναι το μόνο εμπόδιο στην πρόσβαση στις αναγκαίες φαρμακευτικές αγωγές. στην πραγματικότητα τα αρμόδια όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης όχι μόνο αδιαφορούν για τις υπερκοστολογήσεις αλλά και προωθούν συνειδητά πολιτικές περιορισμών στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. στη χειρότερη κατάσταση από όλους βρίσκονται οι χώρες κάτω από καθεστώς μνημονίου όπου η τρόικα ακολουθεί πολιτικές βίαιης πτωχοποίησης με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αδυνατούν να καταβάλουν τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη και να αυξάνεται η θνησιμότητα. στην ελλάδα οι θάνατοι από 108.000 το 2009 αυξήθηκαν στις 117.000 το 2012 ως αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της εγκληματικής πολιτικής της τρόικας. η ευρωπαϊκή επιτροπή Ευχαριστώ κύριε Χρυσόγωνα. Για δύο λεπτά η κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας άκουσα, κυρία Επίτροπε. Αλλά δεν με πείθετε. Διότι 15 κράτη που ε, απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το φως που πήρε αυτό το φάρμακο κατά της πατήτητας γάμα ε, θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι πρόκειται και 50 με 60.000 ευρώ το, για τον κάθε ασθενή, για μερικές εβδομάδες θεραπεία. Ε, θεραπεία που έχει να κάνει με 8, που αφορά μάλλον 8 εκατομμύρια ε, ασθενείς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό όμως το φαινόμενο δεν αφορά μόνο πλέον το συγκεκριμένο φάρμακο, τη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, αλλά μια σειρά από φάρμακα, αντικαρκυνικά και το καθεξής. Και έτσι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα συστήματα υγείας ε, κάνουν ένα εξορθομολογισμό λέγοντας ότι αν κανείς είναι πολύ ηλικιωμένος σε παραδείγματι δεν χρειάζεται τη θεραπεία γιατί τους άλλους δεν θα έχει ε, τη χρησιμότητά της η δαπάνη. Και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα υπάρχει και το πρόβλημα του μονοπωλίου και του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Εάν το διπλώμα ε, ευρεσιτεχνίας έχει διάρκεια 20 ετών υπάρχει ε, λύση από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται τα κράτη-μέλη, δηλαδή υποχρεωτική άδεια που μπορεί να επιβάλλει ένα κράτος και άρα μπορεί να ανοίξει ως εκ τούτου η αγορά και ένα εργαστήριο να αρχίσει να παράγει τα φάρμακα αυτά με πολύ χαμηλότερο κόστο. Η έρευνα επίση, για κοιτάξτε λίγο τι συνέβη με τον έμπολα. Η κρίση που βλέπουμε στην ε, Δυτική Αφρική. Από το 1976 είναι γνωστό ο ιό έμπολα, αλλά κανένα φαρμακευτικό εργαστήριο δεν ε, θέλει να ασχοληθεί και να κάνει είτε θεραπευτικέ αγωγέ, είτε εμβόλια, γιατί δεν είναι οικονομικά ικανοποιητική ή ανταπόδοση. Χρειάζεται λοιπόν δημόσιο χρήμα και εφόσον δίνεται δημόσιο χρήμα πρέπει να δίδεται με όρο ότι δεν θα επικρατήσει μονοπωλιακή κατάσταση ούτε διπλωμαύρη τεχνία. Και άρα θα έχει ο καθένα τη δυνατότητα τη πρόσβαση στο φάρμακο, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και την υποστήριξη κοινοτομία, γιατί έχουμε έλλειμμα κοινοτομία. Ευχαριστώ κύριε Ρίβαση. Κύριο Σταμπουρρόνο, για ένα λεπτό. Χαίρετε είναι ιδιαίτερη ευχαριστησία μου για αυτή τη συζήτηση, γιατί είμαι οδοντίατρος και γνωρίζω τα δράμα της υπατήτητας γάμα και επίσης γιατί εμείς στο κίνημα Τσίνκου Στέλε πιστεύουμε ότι πραγματικά ο φαρμακευτικός ε, κλάδος ε, ε, δεν θα έπρεπε να υπερνικά στην πρόσβαση τα φάρμακα. Θα πρέπει σε κάθε χώρα μέλος να είναι αρμόδιος ο Υπουργό Υγεία. Πώ είναι δυνατόν όταν θα είναι εμπορικοί κλάδοι αυτοί οι οποίοι θα έχουν αρμοδιότητα και όχι ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την προστασία τη δημόσια υγεία. Πώ είναι δυνατόν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στο ε, επιπλέον έχει και καθολική ε, πλειοψηφία όπου προτείνεται ότι θα πρέπει να προστατεύεται η ζωή, να μην μειώνει σημαντικά τις τιμές των φαρμάκων. Σήμερα αρκετέ μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, μου έστειλαν επιστολέ για το, για το θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει να προστατεύσουμε πρωτίστω τη ζωή των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Ταμπουράνο. Για 1,5 λεπτό η κυρία Καϊλή καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα για ρύθμιση των τιμών των παντεντών στα φάρμακα και θα προσπαθήσω να βρω τρόπους να σας διευκολύνω για άλλες λύσεις καθώς η συμφωνία η trips επιτρέπει σε περιπτώσεις φαρμάκων την αδειοδότηση των γενοσύμων εκεί λοιπόν που τα ανθρώπινα δικαιώματα υπερέχουν των πνευματικών δικαιωμάτων και αναρωτιέμαι ενεργοποιήθηκε κατά περίπτωση η γερμανία και η ιταλία γιατί δεν ελέγχεται τουλάχιστον με υποχρεωτική διαφάνεια το πραγματικό κόστος έρευνας των πολυεθνικών και στη συνέχεια σε περιπτώσεις χροκέρδειας να λήγουν στις περιπτώσεις φαρμάκων σε λιγότερο από είκοσι χρόνια οι πατέντες ή να εξορθολογίζονται οι τιμές καθώς θα μπορούσε η ευρωπαϊκή ένωση να αρνείται σε συνεννόηση φυσικά με τα κράτη μέλη μέσω του δημοσίου συστήματος υγείας να παραλαμβάνει και να αγοράζει ε, σε εξωφρενικά ακριβές τιμές τα φάρμακα αυτά. θα μπορούσε λοιπόν να διοδοτήσει γενώσιμα στις περιπτώσεις αισχροκέρδειας ή σε περιπτώσεις που υπάρχει ε, ανάγκη μεγάλη για την υγεία των ανθρώπων. σας ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την ανθρώπινη ζωή είναι μεν πολύ δαπανηρή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παρέχονται φάρμακα στους ασθενείς. Κάθε ασθενή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει ισότιμη ε, διανομή φαρμάκων μεταξύ των ασθενών. Δεν είναι δυνατόν τα φάρμακα αυτά να είναι διαθέσιμα μόνο για τους πλουσίους και όχι για τους φτωχούς, γιατί αυτό αφήνει περιθώριο για όλες αυτές τις πρακτικές τις οποίες θέλουμε να καταπολεμήσουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε πρόσβαση σε φάρμακα, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή η πρόσβαση μόνο σε περιπτώσεις τις οποίες ε, ε πάσει κάποιος από θανατοφόρο ασθένεια. Υπάρχουν και άλλες μορφές παροχής ε, ε, φροντίδας και θεραπείας. Θα πρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς καλής ποιότητας παροχές. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι έχει οριμάσει ε, ο πολιτισμός μας σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούμε να φροντίζουμε τους ασθενείς μας. Δεν είναι δυνατόν ο πολιτισμός μας τη σήμερα ημέρα, αντί να φροντίζει αυτούς οι οποίους έχουν ανάγκη, τους πιο ευάλωτους, να μην επιτρέπει να προσφέρεται η κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη. όλοι τώρα προσπαθούν να βρουν ένα φθηνό τρόπο και προσπαθούν όλοι να εγκαταλείψουν τον κόσμο αυτό μέσω αυθανεσίας, γιατί αυτός είναι ο φθηνός τρόπος. Και πραγματικά προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ε, ε, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ορισμένες φορές μου θυμίζει τους αρχαίους καιρούς, όπου οι κοινωνίες προσπαθούσαν να... Ε, μην ε, έχουν ε, ανθρώπους με αναπηρίες ή ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι και τους πετούσαν στον Κιάδα. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι στη Σλοβακία δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Thank you, Chair. In the context of access... Το, στο θέμα αυτό ε, οι ελλείψεις που προκαλούνται ε, για λόγους παραγωγής, ε, προσφοράς αλλά και για λόγους τιμής. Ε, θα ήθελα να συγκεντρωθώ, να επικεντρωθώ στο τελευταίο. Το πρόβλημα αυτό ε, είναι ιδιαίτερα σοβαρό σε χώρες του, στις χώρες του μνημονίου εξαιτίας της συνολικής μείωσης των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η ίδια η Κομισιόν ε, στις, αναχώρες αναχώρα συστάσεις της λέει ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση στο ε, ε, σύστημα υγείας πλήττει, πλήττουν ε, περισσότερο τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Στην Ιρλανδία αν μεταξύ του 2011 καταγράφηκε μια μείωση στις ε, φαρμακευτικές κατά 17% και ε, από τότε επιπλέον 5%. Ε, αυτό είναι το 1 τέταρτο περίπου ε, του συνολικού μας προπολογισμού. Είναι μεγάλη μείωση. Μετά, διάφορες οργανώσεις και πλατφόρμες των πολιτών ζητούν να, να απαιτήσουμε από τον Επίτροπο να ξαναδεί το θέμα ε, της ε, συμπερίληψης ε, των φαρμάκων και των ιατροφαρμακευτικών συσκευών στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρκιν. Για ένα λεπτό η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, μια φαρμακευτική εταιρεία που ζητάει 50 60 ευρώ για μια θεραπεία ε, τριών μηνών ε, είναι ντροπή. Αν εφαρμοζόταν αυτό στην Πορτογαλία για όλους τους ασθενείς τη C θα έπρεπε να πληρώσουμε ένα ποσό ίσο με το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνη σε όλα τα νοσοκομεία μας. Ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και, η, ε, και τα μονοπόλια αυτή τη στιγμή ε, καταστρέφουν τα συστήματα υγεία μας, υγείας μας. Δεν πρόκειται για καινοτομία. Μόνο το 10% της τιμής ενός φαρμάκου πηγαίνει στην έρευνα. Δεν πρόκειται για καινοτομία, πρόκειται για, ένα, για ένα πρόκειται για το κέρδος και μόνο. Και οι φορολογούμενοι πληρώνουν το υπόλοιπο 90%. Αυτό το κέρδος δηλαδή. Η Κομισιόν λέει δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε σχέση με τις τιμές. Ναι, έχετε πράγματα. Μπορεί να μην μπορείτε να κάνετε κάτι για τις τιμές, αλλά έχετε να κάνετε για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Μπορείτε να καταπολεμήσετε αυτά τα μονοπόλια τα οποία τα χρηματοδοτούν τα κράτη. Μπορείτε να πολεμήσετε αντίον των μονοπωλίων αν έχετε πολιτική βούληση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματίας. Η κυρία Άουκεν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή αποδεικνύει ότι οφείλουμε να αναλάβουμε δράση. Αν η κερδοσκοπία και η αγάπη για το κέρδος της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι τόσο ε, ανεξέλεγκτη, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Έχουμε να κάνουμε με ποσά για την έρευνα και την τεχνολογία που δαπανάει το δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία τελικά μπαίνουν στις έπες της φαρμακοβιομηχανίας. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς ε, διαμορφώνεται όλο αυτό το σύστημα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τους ε, πολίτες να πεθαίνουν. Χρειάζεται η πολιτική βούληση εκείνη. της αντιμετώπισης του φαινομένου που έχει χαρακτηριστεί ως ιδιωτικοποίηση του κινδύνου του κοινωνικοποίηση του κινδύνου και ιδιωτικοποίηση του κέρδου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άουκεν. Για ένα λεπτό κύριο Χρωματικάκης. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα. Εκεί οδήγησε ένα εκρηκτικό μείγμα παραγόντων άμεσα σχετιζομένων με την οικονομική κρίση και τα σκληρά και παράλογα μνημόνια που έχουν επιβληθεί στη χώρα στο πλαίσιο εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης οι τιμές των φαρμάκων μειώθηκαν αισθητά δημιούργησαν όμως παράλληλα σημαντικές παρενέργειες. διάφορες φαρμακοβιομηχανίες μείωσαν τις ποσότητες εισαγωγών ή και τις σταμάτησαν ολοκληρωτικά. οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης όπου οι τιμές είναι υψηλότερες ανάγκασαν τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων να προχωρήσει σε μια σειρά απαγορεύσεων. Μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα δεν έχει τα μέσα να αντισταθεί στην πάυση μείωση εισαγωγών των φαρμακοβιομηχανιών. Είναι λοιπόν απαραίτητο ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα θεσπίσει την υποχρέωση των εταιριών να παρέχουν τα προϊόντα τους και στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες όταν απειλείται η υγεία συμπολιτών μας δεν να καθυστερήσεις που Σας ευχαριστώ κύριε Γραμματικάκη. Για ένα λεπτό η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, τα φάρμακα είναι ε, το τρίτο αίτιο θανάτου μετά τον καρκίνο και τα καρδιακιά νοσήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν γενικευμένες παροχές φαρμάκων. 100 ε, ε, εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν από επίπεδα γάμα ε, παγκοσμίω και 800 περίπου χιλιάδες στην Ισπανία. Πολλοί δεν μπορούν να λάβουν φαρμακευτική αγωγή γιατί δεν μπορούν ε, ε, να λάβουν τα φάρμακα τα οποία προβλέπονται. Υπάρχει μια νέα θεραπεία η οποία μπορεί να βελτιώσει σε 90% την πάθηση αλλά η τιμή της είναι πάρα πολύ αυξημένη και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση σε αυτή τη φαρμακευτική αγωγή από, για την πλειονότητα των ασθενών και φυσικά δεν μπορεί να τα καλύψουν και τα δημόσια συστήματα υγείας γιατί πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ ε, άσχημο να υπάρχουν τόσο υψηλέ τιμέ ε, για φάρμακα τα οποία είναι τόσο απαραίτητα. Ζητούμε μείωση των τιμών αυτών των φαρμάκων που επιτρέπουν ε, την καλύτερη θεραπεία. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την επιδείνωση τη κατάσταση και το θάνατο αυτών των ανθρώπων όταν υπάρχουν θεραπείε οι οποίε είναι αποτελεσματικέ και μπορούν να επιφέρουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Καμπεθόν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε πριν από κάποιους μήνες το σοφοσμπουμπίρ, το οποίο ε, στο 90% των περιπτώσεων θεραπεύει την υπαδίτητα γάβα ε, μέσω αυτής της φαρμακευτικής αγωγής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να διερευνήσει κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα ε, κατάχρησης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που παράγει το φάρμακο συνεργάζεται με την Ινδία και επιχειρήσεις εκεί για να παράγει σε πολύ χαμηλότερη τιμή το γενώσιμο φάρμακο. Πρέπει να γίνει η απαραίτητη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τη διαφάνεια και την ρύθμιση των τιμών των φαρμάκων και των αποζημιώσεων. Ε, θα πρέπει να υπάρχει εξομοίωση των διαφόρων ε, ε, συστημάτων υγείας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διακρίσεις για πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία σώζουν ζωές, όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, πρόκειται για εσωτερική αγορά και είναι αρμοδιότητα και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να γίνονται τέτοια παιχνίδια με την υγεία των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπέσον Ρουίς. Έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των εγκεκριμένων ομιλητών. Έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Με μία παρεμβάση τον κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Επιτροπή μας κάνει μια δήλωση για την πρόσβαση σε ζωτική σημασία σε φάρμακα στην Ευρώπη. Ε, εύκολο είναι να κάνουμε τέτοιου είδου δηλώσεις. Και λέει η Κομισιόν, ανησυχεί για την δυσκολία στην πρόσβαση και για τις τιμές. Για την ανισότητα στην πρόσβαση και θέλει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Η ίδια αυτή η Επιτροπή που, είναι που συμμετέχει στην Τρόικα. Η Τρόικα που στην Πορτογαλία επέβαλε την αύξηση της τιμής των φαρμάκων και την μείωση της ε, συμμετοχής του κράτους. Αυτό οδήγησε σε μείωση της ε, ε, δυνατότητας πρόσβασης. Αυτή τη στιγμή οι χαμηλομισθοί και οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν μπορούν να βρουν φάρμακα ούτε στα φαρμακεία. Τα φαρμακεία που βρίσκονται στα νοσοκομεία δεν παρέχουν φάρμακα. Ε, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα, αλλά είναι υπεύθυνη και η Κομισιόν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι, τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολυεθνικές εταιρείε φαρμάκων, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε στη δράση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερέρα. Έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία Καριστιά και για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα λάβει το λόγο για άλλη μια φορά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος Έντεκαρτ. Ε, καταλαβαίνετε γιατί επειδή είναι αργά δεν πρόκειται να απαντήσω λεπτομερώς. Καταλαβαίνω βέβαια τι εννοείται και θα ενημερώσω τον Επίτροπο Μπόρτς που έχει το θέμα αυτό στο χαρτοφυλάκιό του. Επίσης είναι εδώ οι συνεργάτες του που άκουσαν τη συζήτηση, ε, κράτησαν σημειώσεις και αύριο ήδη οι εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίας ε, εμπειρογνώμες από τα κράτη-μέλη θα συναντηθούν για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Θα είναι λοιπόν μια ευκαιρία και για τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν αυτή τη συζήτηση. Αλλά να πω στον κύριο Φερέιρα που μίλησε για την τιμή των φαρμάκων θα ξαναπώ ότι οι τιμές των φαρμάκων δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, ανταλλαγή πληροφοριών και από όσο γνωρίζω το άτυπο Συμβούλιο Υγείας ε, έχει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξή του στην επόμενη συνάντησή του. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις απόψεις σας. Ε, θα φτάσουν στον Επίτροπο Μπόρτς. Σας ευχαριστώ κυρία Έδικαρτ. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση και η ημερήσια διάταξη για τη σημερινή συνεδρίαση, η αυριανή συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο στις 17 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχετε ε, λοιπόν το ελεύθερο τώρα να επιστρέψετε στα ξενοδοχεία σας για να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ.